συνεχίζουμε την ε, συζήτησή μα. Ε, θα μιλήσουμε για την έκθεση, θα συζητήσουμε την έκθεση πρόσβαση των φορολογικών αρχών στι πληροφορίε για την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εισόδων από παράνομε δραστηριότητε. Έκθεση Μορέλ. Θα δώσω το λόγο για